μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου την Τετάρτη, σύμφωνα με το άρθρο 74 ε, του κανονισμού. Και αυτά θα δημοσιευθούν στα πρακτικά. Πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη, ζητάει το λόγο ο κύριος Γλέζος, παρακαλώ, για διαδικαστικό. Καλό αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι για το εξής γεγονός ότι στην Ελλάδα στις 25 Ιανουαρίου ο ελληνικός λαός εξέλεξε μια νέα κυβέρνηση και τώρα οι δανειστές της εξακολουθούν και επιμένουν να την στραγγαλίσουν. Απευθύνω έκκληση, έκκληση προς όλους να βοηθήσετε να σταματήσει ο στραγγαλισμός του ελληνικού λαού, να μείνει ελεύθερος ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για την τύχη του. Αυτό είναι το αίτημά μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλέσο. Ερχόμαστε ε, τώρα στη διάταξη των εργασιών. Και εσείς για διαδικαστικό, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πριν από δύο εβδομάδες ακούσαμε μια δήλωση για ξενόφοβες και ρατσιστικές δηλώσεις που έγιναν εις βάρος ε, Ρουμάνων και ο Τζανλούκα Μπονάνο ευθύνεται για τέτοιες ρατσιστικές ε, ε, δηλώσεις. Είχε πει ότι οι Ρουμάνοι είναι ικανοί να σκοτώσουν για λίγα ευρώ. Είναι πολύ σοβαρό ένας ευρωβουλευτής να κάνει τέτοιες δημόσιες δηλώσεις και μάλιστα η αποδοχή τέτοιων ισχυρισμών χωρίς τιμωρία δημιουργεί πολύ κακό προηγούμενο και αμαυρώνει την έγκλη και την εικόνα του δημοκρατικού αυτοθεσμικού οργάνου. Θα ήθελα λοιπόν να λάβετε ξεκάθαρη θέση και να επιβάλλετε κυρώσεις στον κύριο Τζαλούκα Μπονάνο για τις ξενόφοβες και ρατσιστικές του δηλώσεις. Και δεδομένων των γεγονότων των τελευταίων δύο εβδομάδων, καλό θα ήταν να γίνει και συζήτηση για το θέμα αυτό. Ε, παρακαλώ. Συνάδελφοι. Ούτε Κανένα από τα προηγούμενα διαδικαστικά δεν ήταν πραγματικά διαδικαστικά. Ήταν ομιλίε επί τη ουσία. Παρακαλώ, όταν ζητάτε το λόγο για διαδικαστικό, να θέτετε διαδικαστικό. Αλλιώ θα μπορούμε να το χειριστούμε όλοι, να το χρησιμοποιήσουμε ω πρόσχημα για να κάνουμε λογίδρια όποτε μα κατέβει. Και αυτό που είπατε δεν ήταν διαδικαστικό ούτε αυτό. Αγαπητή κυρία συνάδελφε Ταπαντέλ, δηλώσεις βουλευτών που γίνονται εκτός του ημικυκλίου και σε αυτό δεν αναφερθήκατε, σε κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κύριος όχι εντός εθούσης, αλλά σε μια συνέντευξη που έδωσε στην Ιταλία. Ε, ε, Λυπάμαι λοιπόν, πάρα πολύ, αλλά δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να δώσω συνέχεια σε αυτό μιλήσατε για τον κύριο Μπουονάνο. Για όλες τις πράξεις και τις δηλώσεις του εδώ στο Κοινοβούλιο είμαι αρμόδιος. Αύριο θα ενημερώσω το Κοινοβούλιο για τις ρυθμίσεις και τα μέτρα που έλαβα κατά τον κύριο Μπουονάνο για πράγματα που διέπραξε εδώ στο Κοινοβούλιο. Κατά τα άλλα, όταν έχουμε δηλώσεις ρατσιστικές, ξενόφοβες και τα λοιπά και άλλες παραβιάσεις, σας παραπέμπω στη δικαιοσύνη της εκάστοτε χώρας. Εγώ εκτός του Κοινοβουλίου δεν έχω την παραμικρή δυνατότητα επιβολής κυρώσεων ή λήψης άλλων μέτρων. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στη διάταξη των εργασιών.